Συνεχίζουμε με τις εργασίες μας, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα δώσω το λόγο στην Μόνικα Χολμάιερ. Θα μας παρουσιάσει ε, το θέμα της σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων. Την αντικαθιστάτε, κύριε Φερνάντη, σωστά. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και θα μιλήσω πορτογαλικά. Η κυρία Χολμαγέρ ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρούσα, γιατί ήταν αδύνατο και εγώ θα κάνω την παρουσίαση εξ ονόματός της. Πρόκειται για την πρόταση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων μέσω χρηματοδοτική στήριξης για τη διαχείριση συνόρων και θεωρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θέτει ένα ανώτατο όριο που πρέπει να πρέπει να γίνει σεβαστό για τις νέες προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα. Εμείς πρέπει να έχουμε πρόσθετους πόρους. Και αυτό φυσικά έχει νόημα. Επομένως, εφόσον έχουμε νέες ανάγκες, θα πρέπει να έχουμε όλο ένα και περισσότερα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, δεν ε, θα πρέπει να έχουμε περικοπές εις βάρος των προγραμμάτων που έχουν δείξει επιτυχία. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε μια ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση αυτή. Και τα ποσά αναφέρονται στην έκθεση. Ακολουθούμε εδώ και την απόφαση της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών σε τρεχούμενες τιμές. Επίσης, έχουμε αυτά τα δύο μέσα που συμπεριλαμβάνονται στο Ταμείο Έχουμε και το θέμα των εξοπλισμών ε, και το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων. Η κυρία Χολμάιερ έχει καταθέσει 14 τροπολογίες. Όπως ήδη σας είπα, είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της Κομισιόν. Είναι θετική πρόταση. Και η συγγήτρια αναφέρει ότι θα πρέπει να μάθουμε από κάποια δραματικά διδάγματα και από τις παρελθούσες εμπειρίες. Διαφάνεια είναι απαραίτητη, η ικανότητα πρόβλεψης είναι απαραίτητη. Θα πρέπει η Κομισιόν να βοηθήσει τα κρατημέλη. για να συμμετέχουν στην επίτευξη του στόχου. Αυτή είναι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σας είπα, απαιτούνται πρόσθετοι πόροι, αλλά και πόροι που να τους διαχειριζόμαστε με διαφάνεια, χωρίς γραφειοκρατία. Η απλούστευση είναι ζωτική και για το στόχο αυτό και για αυτά τα νέα καθήκοντα, για αυτούς τους νέους στόχους, πέρα από τους πρόσθετους ε, πόρους, πρέπει οι πόροι αυτοί να είναι και επαρκής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Χωσέ Μανουέλ, για την παρουσίαση αυτή. Μας παρουσίασε στην γνωματότηση της κυρίας Χολμάγερ. Ποιος θέλει το λόγο τώρα. Κανείς. Κύριος ε, κυρία Ζαλπαντάρ, όχι. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν ε, αντιδράσεις, άρα συμφωνούν όλοι με τα όσα μας είπε ο κύριος Φερνάντες. Δεν έχετε τίποτα να προσθέσετε φαντάζομαι. Ελήψη ανταλλαγή απόψεων. Τώρα, ο κύριος Κύρτσος θα έρθει φαντάζομαι. Ίσως. Οπότε, τότε ο Αλένα Μασούρ να μας παρουσιάσει τη δικιά του γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Άμυνας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, εγώ είμαι εδώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητήθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να γνωμοδοτήσει για τον κανονισμό ε, για τον οποίο επί της ουσίας ε, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ήτρε. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών λοιπόν έχει παρακολουθήσει από την αρχή αυτή την υπόθεση και απεφάνθη σχετικά με δύο δράσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και εφαρμόζονται. Η πρώτη είναι η προπαρασκευαστική για την έρευνα όσον αφορά την άμυνα, γιατί θα θυμόσαστε ότι πρόκειται για 90 εκατομμύρια σε τρία χρόνια. 25 έχουν ήδη δοθεί για το 2017, για τη χρονιά που πέρασε και η πρώτη προσφορά ε, ζητήθηκε για συμφωνίες που θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2018. Και έπειτα από την άλλη υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας βάσει της έκθεσης της Φρανσουάζ Γκροστέτ. Ο στόχος είναι να υπάρξει πρόγραμμα διετές, 2019-2020 δηλαδή, για να στηρίξουμε όχι πια την έρευνα, αλλά την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας. Με 500 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια. Έχουμε ένα σχέδιο κανονισμού λοιπόν που θα ισχύσει στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή μετά το 2020, για 7 χρόνια. Και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ουσιαστικά θα συγχωνεύσει και θα ενισχύσει τις δύο δράσεις που σας ανέφερα τώρα. Με ένα σκέλος που είναι η έρευνα, με ενίσχυση της χρηματοδότησης και ένα σκέλος ικανότητα και πρόκειται για αναπτυξιακά βιομηχανικά προγράμματα. Το Ταμείο αυτό θα έχει 13 δισεκατομμύρια πρικοδότηση για ολόκληρη την περίοδο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου με 5% στις τεχνολογίες ρήξης. Ανατρεπτικές, τις ανατρεπτικές τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβαίνει σε θέματα άμυνας, λοιπόν, και ένα μέρος του προπολογισμού το δίνει και την επόμενη περίοδο θα υπάρξει μια πιο σημαντική διάσταση. με μεγαλύτερη ακόμα σημασία. Όπως προβλέπετε τώρα στον κανονισμό, έτσι θα ενισχυθεί η αυτονομία και η στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, για τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Κομισιόν. Ακριβώς γιατί πρέπει να πρόκειται για την ευρωπαϊκή διάσταση. Πρέπει δηλαδή επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ερευνητές οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι, δεν είναι βασισμένοι στην ευρωπαϊκή επικράτεια, ανεδρεύουν δηλαδή εδώ, για να υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση. Πολλές από τις χώρες μας σήμερα για τον βαρύ πλεισμό τους εξαρτώνται από ξένες χώρες. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή προτίμηση για το στρατιωτικό εξοπλισμό. Επίσης η πρόταση προτείνει και συμφωνώ και με αυτό τα προγράμματα αυτά να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χωρίς περιορισμούς και να βασιζόμαστε στην αρχή της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής απόδοσης. Όσον αφορά το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να Ξέρετε ότι έχω υποβάλει κάπου 12 τροπολογίες για να διευκρινίσω κάποια σημεία και να τροποποιήσω τη διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποια σημεία. Είναι σαφές ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της άμυνας. Κυρίως όταν πρόκειται για την επιλογή το κόστος της επιλογής, το άμεσο και το έμεσο κόστος επίσης. Το έμεσο κόστος διασφαλίζεται, αλλά βάσει συγκεκριμένων λογιστικών στοιχείων που έχουν εγκρίνει οι εθνικές αρχές. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια εναλλακτική λύση στο σύστημα του καταποκοπήν ποσού 25% έτσι όπως προτείνει ο εισηγητής της ΣΥΤΡΕ. Κατά τη γνώμη μου, και θα επανέλθω εδώ, πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Σίγουρα θα υπάρξει ευρεία συνένεση, ώστε όπως προτείνεται στον κανονισμό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παίξουν σημαντικό ρόλο στην χρήση του ταμείου αυτού. Το ζήτημα το πολιτικό που τίθεται είναι πρέπει να υπάρξει θετική διάκριση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορισμένων χωρών. Αυτό που μας ενδιαφέρει στην Ευρώπη είναι η ευρεία κατανομή των δραστηριοτήτων αυτών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως όμως, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Υπάρχει εξυγχρονισμός, εξοπλισμός εχμής. Κάποιες χώρες έχουν την αναγκαία πραγματογνωμοσύνη, οπότε δεν πρέπει να καθυστερήσει ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού βάζοντας κριτήρια που θα οδηγούσαν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Συνεπώς, δεν είμαι κατά του να υπάρχει ένα σύστημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάποιων χωρών. Όμως, προτείνω να ορίσουμε δύο κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα όλες οι μικρομεσαίες, από όποια χώρα και αν προέρχονται. Να έχουν ως πλονέκτημα να μπορούν να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μπόνους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των χωρών που δεν συμμετέχουν στο κοσόρσιουμ της γενικής επιχείρησης η οποία υποφελείται από την συμφωνία αγοράς και που χρησιμοποιεί ως υπεργολαβία άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας συμβιβασμός που θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ένα επιπλέον μπόνους. Εκείνες δηλαδή που είναι από χώρες που δεν διαθέτουν σήμερα μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Επίσης, είμαι υπέρ. Η εποφελούμενοι από τα κονδύλια αυτά να μπορούν εφόσον θέλουν να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον χρηματοπιστωτικά μέσα από το μέσο Invest EU. Δεν βλέπω γιατί όχι. Τέλος, για τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων. Πιστεύω ότι αυτά που προτείνει ο κανονισμός, το σχέδιο κανονισμού. Και ο εισηγητής της ΣΥΤΡΕ δεν φτάνουν. Θα ήθελε ειδική έκθεση του λεκτικού συνεδρίου. Παρουσίαση της έκθεσης αυτής σε εμά και στον έλεγχο προπολογισμού. Να συμπεριληφθεί και αυτό στον κανονισμό, παρακαλώ. Αυτά όσον αφορά τις τροπολογίες που θα προτείνω στην Ήτρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση της έκθεσής σας και για τις τροπολογίες που θέλετε να μας προτείνετε. Θα ήθελα να στραφώ στους σκιώδεις εισηγητές, η κυρία Χόφμαν. Ε, ίσως ε, εκπροσωπείται από την κυρία Τια Σερμπάλ. Ναι, τελευταία στιγμή αρρώστησε και εγώ δεν έχω πολλές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία συμφωνούμε, γιατί ακολουθεί τη γραμμή που συμφωνήσαμε. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο τροπολογίε. Η έκτη που έχει να κάνει με την ε, συμμετοχή των Βρετανικών επιχειρήσεων και η έντεκα που έχει να κάνει με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν μέρο και του InvestEU, όπου θα γίνει μια ει βάθο ε, συζήτηση στην ομάδα μου, κυρίω ό,τι αφορά το InvestEU. Γιατί όταν ε, μιλούσαμε για αυτό το πρόγραμμα, υπήρχαν αρκετές αμφιβολίες για το αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό και για την άμυνα ή όχι. Αυτά μπορώ να πω τη στιγμή, όμως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πάετ ίσω έχει ζητήσει τον κύριο Ντεπρέ. Όχι. Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Κύριε Σιγητά, είπατε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολιτικό πρόγραμμα που θα πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως θα μπορούσαμε μέσω τροπολογιών να συμπεριλάβουμε μία έκκληση κάπως προκλητική, να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να αναρωτηθούν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των ε, δαπανών σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ασφαλεία και την άμυνα. Και ίσως να τους ζητήσουμε να καταλογραφήσουν τις δαπάνες που δεν έχουν πλέον χρησιμότητα και που θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αν ε, κάποια κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, θα μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση του ευρωπαϊκού προπολογισμού, έτσι ώστε να προχωρήσει ο ευρωπαϊκό προπολογισμό και να αυξηθεί χωρί ε, να έχουμε επιβάρυνση. Γιατί θα δείξουμε και ποια είναι και η προσθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, εγώ το χαιρετίζω με ξεπεράσατε. Υπάρχει 10 Οκτωβρίου η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου μπορούμε να δεχτούμε τις τροπολογίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι θετικό να έχουμε μια τέτοια τροπολογία. Γιατί, για την άμυνα. Μια ένα από τα παράδοξα της συζήτησης που είναι τόσο παλιό όσο και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ότι περιοδικά ακούμε διάφορες ε, φωνές ε, που μας αναφέρουν ποιος είναι ο κίνδυνος ε, της επικάλυψης των δεπανών μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτή η καταπληκτική επικάλυψη που υπάρχει σήμερα είναι ότι έχουμε 28 προϋπολογισμούς για την άμυνα, 28 χωρών, που η κάθε μία έχει ένα στρατιωτικό εργαλείο και καμία δεν μπορεί να πει σε τι θα χρησιμεύε σε περίπτωση συγκεκριμένης κρίσης και μάλιστα ακόμη και οι καλύτερα εξοπλισμένες χώρες ε, δεν μπορούν να διεξάγουν αυτό που θα αποκαλούσαμε πόλεμο. Τώρα το αποκαλούμε δράση υψηλής έντασης. Πρόκειται για έναν τομέα όπου έχουμε ε, τεράστιες ε, κρίσεις σε σχέση με την εξοικονόμηση. Εγώ συμφωνώ λοιπόν και με τα τέσσερα χέρια, αν θέλετε, να το γράψουμε, να τη γράψουμε αυτή την πρόταση και μάλιστα και με του συναδέλφου που συμμερίζονται την ανάλυση αυτή. Πρόεδρος, αυτές οι παρεμβάσει υψηλή έντασης, αν μπορούσαν να ανοίξουν ε, ευρέως την πόρτα τη μετανάστευση. Ε, Παραδείγματο χάρη σκέφτομαι ε, τι συνέβη με την Αραβική Άνοιξη, δεν έχουμε πλέον κράτος στη Λιβύη. Οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν αντικαταστήσει το κράτος. Και ο εμφύλιος πόλεμος ε, έχει θέσει κίνηση εκατομμύρια σύρους σε δραματικές συνθήκες. Αν ε, θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να πούμε κάτι για την κατάσταση αυτή, εγώ δεν θα δίσταζα Κύριε Σιγητά, ίσω θα μπορούσαμε να καταθέσουμε μια τροπολογία. Ωραία, Πρόεδρα. Η Επιτροπή Προπολογισμών είναι εντό του ρόλου τη στο να επιμείνει στην ε, καθήλια αρμόδια επιτροπή ότι αυτά τα κονδύλια, αυτό το ταμείο θα πρέπει να συμβάλλει στην εξοικονόμηση και να βελτιώσει τη σχέση κόστους-οφέλους ε, των 28 αμυντικών μας συστημάτων. Πρόεδρος, θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουμε τις τροπολογίες μας μέχρι τις 3 το μεσημέρι στις 10 Οκτωβρίου και αυτό αφορά το σύνολο των τροπολογιών. Η Επιτροπή Προβλησμών θα αποφανθεί στις 5 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Λάμα Σουρ και την ε, κυρία Γκαρσία Σαμπάλ και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κίρτσο. Γεια μέσο για τον ε, τελωνιακό έλεγχο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησής μου της Επιτροπής Προϋπολογισμών αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θεσπίζει στο πλαίσιο του Ταμείου Γενικονοικονομικής Διαχείριση των Συνόρων το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνιακών ελέγχων. Επί της ουσίας αρμόδια η Επιτροπή ΙΜΚΟ εσωτερικής αγοράς, δηλαδή και προστασίας των καταναλωτών. Είναι σύντομη και σχετικά τεχνική γνωμοδότηση. Έχω υποβάλει δύο τροπολογίες. Και ε, ε, η μία αφορά κάποια ειδικά θέματα και το δεύτερο ε, τα θέματα του δημοσιονομικού κανονισμού. Όπως έγινε και σε άλλες νομοδοτήσεις για την περίοδο 21-27, ε, όπως είναι ε, τετελωνία και ε, η υπηρεσία διαστήματος. Τα σημαντικότερα είναι τα οικονομικά στοιχεία, οικονομικός φάκελος για το μέσο αυτό για την περίοδο 21-27 θα είναι 1 δισεκατομμύρια 149 εκατομμύρια, σε τιμές ε, του 2018, δηλαδή ένα δις 300 εκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές. Ε, το ποσό αυτό προτείνεται να ευθυγραμμιστεί ε, με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14 Μαρτίου και 13 Μαΐου ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και αναμένονται και άλλες προσαρμογές όταν έρθει η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνολικό επίπεδο 1,3% του προϋπολογισμού του, 1,3% του ΑΕΠ να είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκτός αυτού θα μπορούσαμε να προτείνουμε και άλλες τροπολογίες έτσι ώστε τα προγράμματα εργασίας να γίνουν από κατεξουδότης πράξης και όχι ε, εφαρμοστικέ. για να έχει λόγο το Κοινοβούλιο. Αυτό ζήτησε και ο συντάκτης νομοδότησης για το ορίζον. Αυτό συνάδει περισσότερο με την πάγια αρχή ε, του Κοινοβουλίου, αλλά είναι μάλλον αρμοδιότητα και εξουσία της ε, αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπή της ΙΜΚΟ να το προτείνει και όχι δική μας. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Και τώρα στρέφουμε προς τους σκιώδησίτες. Η κυρία Χόφμαν, διαστόματος ε, Ίντερ Γκαρδία Σάμπαλ. Όχι. Ο κύριος Αλή, διαστόματος του κυρίου Ντεπχέ. Ούτε εσείς. Θέλετε. Όχι. Νομίζω ότι η σιωπή των σχεδόν ε, ε, εισηγητών είναι προς απάντησή σας κύριε εισηγητά, τα είπατε όλα. Οι τροπολογίες θα πρέπει να καταθεθούν μέχρι τις 2 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και η Επιτροπή μας θα τις εξετάσει και θα αποφανθεί με ψηφοφορία στις 5 Νοεμβρίου. Προχωρούμε. Θα ακούσουμε τον συνάδελφο Χόβαρτ. Σέσπιση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημιουργική ε, ε, οικονομία καμιά φορά θεωρείται κάτι το, το επιπόλαιο που σου λέει σιγά τι παράγει ο άλλος, δεν έχει οικονομικό ενδιαφέρον, ε, απλώς είναι ένας κλάδος που απομιζά δημόσια κονδύλια. Αυτό είναι τεράστια πλάνη και στρεβλή αντίληψη και γενικά αυτά είναι κάποιες νοοτροπίες ε, της κατασκευαστικής οικονομίας που σνομπάρει τη δημιουργία. Εδώ πρόκειται για κλάδους που παράγουν δισεκατομμύρια και σε παγκόσμιες αγορές και πραγματικά θα πρέπει η ευρωπαϊκή αυτή παραγωγή και δημιουργεί να μπορούν να ανταγωνίζονται σε διεθνές περιβάλλον. Και είναι και πολύ κερδοφόρος αυτός ο κλάδος πολλές φορές με σχολές αριστείας και ιδρύματα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να υποστηρίζονται οικονομικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου χρειάζεται ενίσχυση γιατί ε, ε, υπάρχει και ε, στην επιστήμη, ας πούμε, η βασική έρευνα, η θεμελιώδης και εφαρμοσμένη. αντίστοιχα, χρειάζεται μια υποστηρικτική δράση και η δημιουργία έτσι ώστε να προχωρεί καλύτερα εξού και είναι τόσο πολύτιμο το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. η Δημιουργική Ευρώπη ε, αφορά και τον πολιτισμό και τις παραδόσεις, αλλά μπορεί να έχει και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ε, διαφυλάσσοντας τη γλωσσική ποικιλομορφία ε, και σε αυτό φιλοδοξεί και έχει ρόλο να διδραματίσει το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Στη γνωμοδότησή μας τώρα έχω καταθέσει εγώ 8 τροπολογίες που αντανακλούν τη σημασία των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και τη συνέχεια και τη συνέπεια των ποσών και των ε, αριθμητικών στοιχείων που έχουμε στο PDP στις σταθερές τιμές. Και δύο συγκεκριμένους τομείς θέλω να αναφέρω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η διαφάνεια στην αναφορά των ε, χρηματοδοτήσεων που δίνονται στα προγράμματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τρίτες χώρες. Αυτό είναι ε, ένα στοιχείο που διατρέχει όλη μου τη γνωμοδότηση και έχει σημασία να δούμε τι δίσδυση έχουν τα προγράμματα και πώς χρηματοδοτούνται και πόσο πιάνει τόπο η δική μας χρηματοδότηση. Και σχετικό με το πρόγραμμα αυτό είναι ένα σήμα, μια σφραγίδα αριστείας που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Όπως και σε άλλα προγράμματα, το πρόγραμμα αυτό έχει τρομερή ζήτηση. Ε, τώρα ποιοτικά δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι όλες αυτές οι αιτήσει ε, εύστοχες. Χρειάζεται μια ανάλυση για να δούμε εάν ε, θα μπορεί να απονέμεται αυτή η σφραγίδα το βραβείο ποιότητα, α πούμε, αριστεία σε προγράμματα που θα άξιζαν χρηματοδότηση, αλλά που για λόγου αμυγό δημοσιονομικού δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Γιατί η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. Και έρχομαι λοιπόν ε, στα οικονομικά. Η σημερινή γνωμοδότηση αναφέρει κάποια οικονομικά στοιχεία από το PDP. Συνεχίζω τις συζητήσεις με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Πολιτισμού και αλλού για ε, το, την τάξη μεγέθους αυτής της χρηματοδότησης και θα σας κάνω και αντίστοιχη τροπολογία. που θα εκφράζει πιο εύστοχα τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Και τέλος, η άμεση χρηματοδότηση του προγράμματος για δύο ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινηματογράφου που κάνει τεράστια δουλειά στην προώθηση του κινηματογράφου και η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πραγματικά ένα άριστο σχήμα μουσικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν Δημιουργική Ευρώπη προβλέπεται άμεση χρηματοδότηση αυτών των δύο θεσμών και όχι δια της εθνικής. Είναι πραγματικά ο κατάλληλος μηχανισμός. Δεν το αναφέρω στις τροπολογίες γιατί δεν υπάρχει λόγος. Απλώς ήθελα να το τονίσω ε, στην αιτιολόγηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Merci, merci, Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Ο κύριος Χρυστοφόρ, καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πολύ εύστοχα όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από τον αγαπητό εισηγητή που ακουμπούν την ε, ουσία του ζητήματο, γιατί όταν μιλάμε για δημιουργική Ευρώπη ουσιαστικά αναφερόμαστε στον ορισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πρωτίστως ε, για τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό τη και μετά και όλα τα άλλα. Και αν σήμερα κρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για του οικονομικού τη δείχτε, για μένα έπρεπε να θεσπιστούν και πολιτιστικοί δείχτε για να δούμε αυτή η Ευρώπη πόσο δημιουργική και πόσο πνευματική και πολιτιστική ανάταση έχει μέσα σε όλη αυτή την πορεία και θεωρώ μάλιστα ότι τα 541 εκατομμύρια που δίνονται ουσιαστικά για την πολιτιστική ανάπτυξη και τον πολιτισμό είναι ελάχιστα με το εύρος και τη διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών, πολιτισμικών, παραδοσιακών αξιών που προβάλλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξορισμού άρα η Ευρώπη είναι πολιτισμός και κάθε ευρώ, και γι' αυτό απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επενδύουμε στον πολιτισμό είναι πολλαπλάσια επένδυση για το παρόν και το μέλλον τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθησαν προηγουμένω οι δράσει τη Δημιουργική Ευρώπη και μέσα σε αυτέ συμπεριλαμβάνονται διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με διάφορα χειρήματα που εγώ τα θεωρώ πολύ αποτελεσματικά και πολύ σημαντικά, ακόμα και τον, στον τομέα των μέσων ενημέρωση. Η Ευρώπη στερεί στο να μπορέσει να προβάλλει και να διαφημίσει το έργο, τι αξίε τη, τι αρχέ τη και ό,τι ο κόσμο θα ήταν πολύ διαφορετικό αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο δεν προβάλλεται αυτό και δεν γίνεται χτήμα των λαών αυτή η σωστή προβολή και διαφήμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί που πραγματοποιούνται εκατοντάδε θετικά ζητήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Κοσμογονία, οι πάντε ε, ουσιαστικά προπαγανδίζουν και αναβαθμίζουν και φουσκώνουν το ένα ή το δύο ή τα τρία αρνητικά που μπορεί να επισυμβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και ο τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι σημαντικό όπλο στη σύγχρονη εποχή μα να στηρίξουμε τα μέσα ενημέρωση σε όλε τι χώρε για να μπορέσουν να προβάλλουν αυτό το οποίο συμβαίνει, την πραγματικότητα. Και όχι να προβάλλονται τα fake news ή όλα τα άλλα που στρεβλώνουν την πραγματική εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε όμω να πω ότι η απαφορμή αυτού του γεγονότο, παρά το ότι δεν είναι αυστηρά μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματο τη Δημιουργική Ευρώπη, για τον πολιτισμό να πω ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα μέσα σε αυτά τα πλαίσια για να διαφυλάπτει και να προστατεύει τους πολιτιστικούς θησαυρού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον τρίτο χώρο. Εδώ στην Ευρώπη καθημερινά καταστρέφονται πολιτισμοί χιλιάδων χρόνων. Στην πατρίδα μου την Κύπρο καταστράφηκε πλήρως ένας πολιτισμός ελληνοχριστιανικός για χιλιάδων χρόνων. Πλήρω και δεν δόθηκε ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει αυτός ο πολιτισμός να αναστηλωθεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε καταστρέφεται πλήρω ο χριστιανικός πολιτισμός της Μέση Ανατολή. Μέσα από την οργιώδη επέλαση των ακραίων ε, ομάδων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν και δεν είναι παρούσα. Εμείς θα θέλαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντανακλά τη δράση τη πρωτίστω και σε αυτά τα ζητήματα. Είναι εκεί που παίρνει αξία και πιστεύω ότι αν απευθυνθούμε στου Ευρωπαίου που καταβάλουν ουσιαστικά από το ειστέρημά του τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ρωτήσουμε αν αυτά τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτού του σκοπού, είμαι βέβαιο ότι θα απαντήσουν με συντριπτική πλειοψηφία ότι πρέπει να πάνε για να προστατεύσουν τον χριστιανικό πολιτισμό τη Ευρώπη που καταστρέφεται εντό Ευρώπη και εκτό Ευρώπη. Εάν ταυτόχρονα του ρωτήσουμε αν πρέπει να δίνουμε λεφτά σε αυτού που καταστρέφουν τον πολιτισμό, οι πάντε θα μα έλεγαν δεν πρέπει να δίνουμε ούτε μία. Δυστυχώ υπάρχει μια χώρα που καταστρέφει όχι μόνο τον πολιτισμό τη πατρίδα μα, τον ελληνοχριστιανικό, αλλά και του πολιτισμού των γύρω χωρών που εισβάλλει, που είναι η Τουρκία και αυτή η Ένωση Ευρωπαϊκή συνεχίζει να την χρηματοδοτεί. Και θεωρώ ότι χρηματοδοτεί και για τον πολιτισμό αυτή τη χώρα. Και αν ρωτήσουμε του Ευρωπαίου πολίτε σήμερα τι 500 εκατομμύρια, αν πρέπει να χρηματοδοτείται αυτή η χώρα, όλοι θα μα πούν ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτείται. Και αν εμεί παίρνουμε αποφάσει και βάλουμε κυρώσει για χώρε ακόμα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και καλά πράττουμε, πέστε μου ποια κύρωση επιβλήθηκε σε αυτήν τη συγκεκριμένη χώρα. Με αυτά όλα θέλω να πω ότι οφείλουμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό. Το 1 δισεκατομμύριο 850 εκατομμύρια πιστεύω ότι είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, παρά το ότι είναι σημαντικό ποσό, σε αυτό που εμεί έχουμε ενώσει ιδεολογία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι Ευρωπαϊκέ Αρχές και Αξίε. Στηρίζουμε το πρόγραμμα, σε μεγάλο βαθμό στηρίζω και τι τροπολογίε του αγαπητού συναδέλφου και τον συγχαίρω για την εκπληκτική ε, δουλειά και την επικέντρωσή του στην ουσία του ζητήματο για μια πραγματικά πολιτιστική, δημιουργική Ευρώπη που να αντανακλά και την ιστορία και το παρελθόν τη αλλά και το μέλλον της. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι το έτος 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ίσως είναι πιο εύκολο να λέμε ότι είναι το 2018 αυτό το έτος παρά να εγγράφουμε σημαντικές πιστώσεις στον προπολογισμό. Η κυρία Σατερμάκη. κυρία Γιατεμάκη νομίζω έχει εξουδετήσει στον κύριο Ντεπρέ. Μάλιστα, σωστά τα είπατε, Πρόεδρε. Θέλω να πω στον εισηγητή ότι διάβασα την πρόταση του στο εκτιμώντας 18 και στο άρθρο 7 παράγραφος 3 σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα να δημοσιεύονται οι συνεισφορές των τρίτων χωρών στο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι είναι μια λογική πρόταση, όμως έχω μια ερώτηση για όλες τις συνεισφορές των τρίτων χωρών στα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή δημοσιεύει, ίσως να μην το γνωρίζω, ένα συνθετικό έγγραφο που μπορούμε να δούμε για όλα τα προγράμματα της Ένωσης, δηλαδή να έχουμε τις συνεισφορές των διάφορων τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες χώρες σε ορισμένα προγράμματα. Υπάρχει κάποιο τέτοιο γενικό έγγραφο. Υπάρχει κάποιο που θα μπορούσα να το βρω και μου έχει διαφυγεί. Να θέσω μια συμπληρωματική ερώτηση σε αυτή του κυρίου Ντεπρέ. Και αν υπάρχουν ε, συνεισφορές από τις τρίτες χώρες, αυτές ε, αφαιρούνται από τις πιστώσεις που δεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή είναι πόροι που ε, είναι εντός ή εκτός προϋπολογισμού. Ο κύριος Ράιλ. Ευχαριστώ για την ερώτηση, Πρόεδρε και κύριε Ντεπρέ. Σε ό,τι φορά την ερώτηση του κυρίου Ντεπρέ, θα πρέπει να ενημερωθώ δεν ε, βλέπω να υπάρχει συγκεκριμένη έκθεση που να μας δίνει μια καθολική εικόνα των ε, συνεισφορών των τρίτων χωρών, όμως θα στείλω γραπτό στην απάντηση πολύ γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση του Πρόεδρου, η συνεισφορά των τριών χωρών πρόκειται για έσοδα ε, που προστίθεται στις πιστώσεις που έχουν ψηφίσει οι δημοσιονομικές αρχές. Έτσι λοιπόν είναι εκτός ε, ε, του δημοσιονομικού πλαισίου και είναι εκτός του ανώτατου ορίου. Αυτή η διαδικασία που θεωρώ ότι είναι αντίθετη με τις θεμελιώδεις αρχές του προϋπολογισμού η αρχή της καθολικότητας, δηλαδή θα πρέπει όλα τα έσοδα να χρηματοδοτούν όλες τις δαπάνες. Ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν σέβεται τις ίδιες τις αρχές του. Θα μου πείτε δεν είναι σοβαρό γιατί δεν σέβεται καμία αρχή. Δεν σέβεται την ενότητα του προπολογισμού, ούτε την καθολικότητα, ούτε τον ετήσιο χαρακτήρα και αμφιβάλλω αν σέβεται και την ειλικρίνεια. Αλλά, ειλικρινά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που δίνει συμβουλές σε όλους και σε κάθε, κράτη σε κάθε το βρίσκω απαράδεκτο να γίνεται αυτό. Κύριε Δεπρέ, μια διευκρίνηση. Όταν ε, είπατε ότι είναι ε, έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί, δηλαδή δεν μπαίνουν στον προϋπολογισμό, στον νότατα αόρια ε, του πολιτικού προγραμματισμού, αλλά μπαίνουν μέσα στον ετήσιο προϋπολογισμό. Πώς γίνεται με τον ετήσιο προϋπολογισμό δεν εμφανίζονται στον ετήσιο προπολογισμό. Όχι. Δεν έχουν ψηφιστεί αυτά τα κονδύλια από τις δημοσιονομικές αρχές. Προστίθενται στα κονδύλια που έχουν ψηφιστεί. Περίεργο αυτό. Okay. Θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσω και το μικροφωνό μου. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ. Περίμενα να πλήσετε το θέμα που συζητούσαμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε επί των ε, εισφορών. Αλλά αυτό θα πρέπει να ξέρουμε τουλάχιστον περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να έχουμε διαφάνεια εδώ τι δαπανάτε εντό των προγραμμάτων. Διαφορετικά πώς λαμβάνεις αποφάσεις για τα προγράμματα υποψιάζομαι ότι αυτό θα γίνει πιο εμφανές και αυτός είναι ένας ε, από τους λόγους που τέθησα σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θέτει κάποιο πρόβλημα στο να αντικατοπτρίσει το χριστιανικό πολιτισμό και το τι κάνει είναι ένα σημαντικό σκέλος σκεπτικού στον πολιτιστικό τομέα και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει τον εαυτό του με πολλούς τρόπους. Ε, βέβαια, δεν ε, το βλέπουν όλοι ίσως εκ πρώτης όψεως. Πριν το σχάρι έχουμε τη θρησκευτική μουσική. Πάντως αυτό είναι ουσιαστικό τμήμα του πολιτισμού, είμαι σίγουρος, και θα συνεχίζουμε να λαμβάνουμε στήριξη. Σε ό,τι αφορά την συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα, ε, έχουμε γραφεία του προγράμματος σε διάφορες ε, τρίτε χώρες, Μολδαβία, Λευκορασία, Ισλανδία, δεν ξέρω υπάρχει και στην Τουρκία. Όμω, νομίζω ότι πρέπει να αντικατοπτρίσουμε το γεγονό ότι πολλοί από αυτούς τους πολιτισμούς που γίνονται πολιτισμοί κυρίαρχοι εντός της Ευρώπης ε, έχουν ήδη προωθηθεί σε πολλά μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να δούμε τι χρηματοδοτεί ε, αυτό το πρόγραμμα Σκεφτείτε το εξή. Ο μεγαλύτερος δικαιούχο ε, από το media stream του προγράμματο ε, είναι ε, η αρχή του η αρμόδια αρχή για τον κινηματογράφο και η σχολή κινηματογράφου στη δική μου εκλογική επαρχία. Δηλαδή, ωφελούνται οι φοιτητέ σε 80 90%. Δεν είναι βρετανικό το πρόγραμμα αυτό. Το θέμα βέβαια είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε την χρηματοδότηση κάτι τέτοιου ή αν θέλουμε να επαναφεύρουμε τον τροχό. Όμω ε, ήδη η βιομηχανία του κινηματογράφου, ο κλάδο του κινηματογράφου, επωφελείται από αυτό το πρόγραμμα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανυπομονώ να λάβω και τι ε, τροπολογίε και να περάσουμε και στην ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν στις 9 Οκτωβρίου πριν από τις 6 το απόγευμα και η ψηφοφορία των τροπολογιών θα γίνει στην Επιτροπή μας ε, στις 5 του μηνός. Τώρα περνάμε στον συνάδελφο Πόλο Ρουμπίκ για την ψηφιακή Ευρώπη. Αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ψηφιακή Ευρώπη λοιπόν και το πρόγραμμα θα επηρεάσουν πάρα πολύ την ε, απασχόληση και την πρόοδο του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές ε, στα ποσά. Η θέση του Κοινοβουλίου ε, λήφθη μεν υπόψη, αλλά για καλό και για κακό θελήσαμε να εκφράσουμε τις ε, τιμές, ε, τα ποσά σε σταθερές τιμές του 2018 για να μην υπάρχουν περιθώρια ερμηνεών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τις υποψηφιότητες και τη συμμετοχή στα προγράμματα να είναι εναρμονισμένα όλα αυτά. Γι' αυτό προτείνω να αλλάξει ε, το άρθρο 13 και το άρθρο 20. 21 για ε, τους νέους επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες. Μέχρι τις 28 του μηνός θα έχουμε τις μεταφράσεις, τροπολογίες μέχρι τις 9 Οκτωβρίου και εμείς θα ψηφίσουμε 5 Νοεμβρίου εδώ στην Επιτροπή μας αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το μέλλον μας. Οι σκιώδεις εισηγητές. Ο συνάδελφος Deutsch. Ο κύριος Πόπα. Ο κύριος Τόρβαλτς. Ή ο κύριος Ντεπρέ τότε. Mm. Τίποτα δεν έχει να προσθέσει ο κύριος Ντεπρέ. Υπάρχει η απόλυτη τιποτα δεν απόψεων από ό,τι φαίνεται με τον εισηγητή, τον κύριο Ρούμπικ, σωστά. Λέω ο πρόεδρος. Καλώς, κύριε Ρούμπικ. Νομίζω ότι η σιωπή είναι ενθαρρυντική. Δείγμα σοφίας του Κοινοβουλίου μας. Οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν σε 1 Οκτωβρίου πριν από τις 6 το απόγευμα. Και κύριε Ρουμπίκ, μια που μπήκατε στη διαδικασία θα συνεχίσετε με το πρόγραμμα για την ενία αγορά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτό είναι τώρα ένα πρόγραμμα που αφορά τα δύο τρίτα των εργαζομένων στην Ευρώπη. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα μικρομεσαίων που παράγουν το 50% της ε, υπεραξίας στην Ευρώπη και πληρώνουν το 80% των φόρων που χρειαζόμαστε για την κοινωνική πολιτική. Οπότε η ενίσχυση των μικρομισών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερο μέλημα και αγωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εδώ πάλι τα ποσά είναι σε σταθερές τιμές το 2018, άρα δεν χωράνε ερμηνείες και παρερμηνείες. Σε μια τροπολογία είναι όλα αυτά. Και επίσης ε, πήρα νέες προφορίες ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τμήμα του προπολογισμού που δεν είναι εγγεγραμμένο ε, αλλά αυτό ήρθε μετά τη σύνταξη της νομοδότησης και παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει στο μέλλον. Η συνεργασία μας είναι ε, κρίσιμη. Ε, και γιατί αυτό το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό. για την, τον κατάρτιση και τη διατήρηση των υφισταμένων προγραμμάτων. Και σίγουρα θα κάνουμε και τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Κάτι άλλο που έχει σημασία για μας είναι μια κεντρική ιδέα, μια φράση που έχουμε αποφασίσει εδώ στην Επιτροπή μας και είναι θέμα αρχής για μας. Ο διπλασιασμός των πόρων και διατήρηση της χρηματοδότησης για τα τρέχοντα προγράμματα. Γιατί στο κάτω-κάτω πρόκειται για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει να τονωθεί και να ενισχυθεί. Αυτό έχει να κάνει και με εκπαίδευση και με κατάρτιση και με εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα δίκτυα Enterprise Europe ε, έχει μια πολύ καλή διείσδυση στην Ευρώπη και βοηθάει τις εταιρείες να συμπληρώνουν τις πολύ δύσκολες αιτήσει ε, και βοηθάει γενικότερα και με την ανταλλαγή ε, νέων ε, επιχειρηματιών. Το πρόγραμμα Εράσμους για νέους επιχειρηματίες έγινε μια πρώτη δοκιμή, ε, επέτυχε πάρα πολύ και παγκοσμίω τώρα έχει εκφραστεί ενδιαφέρον τέτοιων ανταλλαγών επιχειρηματιών. Έτσι κι αλλιώς ο έρασμος είναι από τα πιο δημοφιλή προγράμματά μας και τα πιο επιτυχή, ιδιαίτερα για τους νέους. Είναι πολύ ωραίο να γνωρίζουν και άλλους πολιτισμούς. Και οπότε υποστηρίζω ε, τα αιτήματα που έχουμε ήδη εκφράσει. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η, η μετάφραση θα έχει φτάσει μέχρι τις 3 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή της γνωμοδότησής σας. Σκιώδης εισηγητές τώρα. Δεν είναι εδώ ο κύριος Ντόιτς. Εκ μέρους του ΕΛΚ. Ο κύριος Ουρίγκα έτσι κι αλλιώς. Καλύπτηκε η κύριε Γαζδαμπάλ όμως. Αυτή τη φορά είσαστε εσείς κοιόδης συζητήτρια. Ναι, Ευχαριστώ. Συμφωνούμε με τη γραμμή του κύριου Ρουμπίκ. Αυτό που δεν έχω καταλάβει καλά, γιατί κατάλαβα το πρόβλημα με τα νούμερα και την συνομιλία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αλλαγή, τέλο πάντων ότι υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε λυθεί υπόψη και ο κύριος Ρουμπίκ το λάβανε υπόψη. Θέλω να ξέρω, θα τροποποιηθούν τα νούμερα για να συνεχιστεί ένα μέρος του προγράμματος να μην περιλαμβάνεται ή όχι. Θέλω να μου το εξηγήσει αυτό κύριο Ρουμπίκ. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε. Ευχαριστούμε κύριε Καρτεσταμπάλα. Η κυρία Ετοιμάκη σας έχει αφήσει κάποιο μήνυμα για μας, κύριε Ντεπρέ. Ναι, ακριβώς. Μου ανέθεσε εντολή. Λοιπόν, τι λέει. Λέει ότι ευχαριστεί τον κύριο Ρούμπικ. Ξέρετε και όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την ομάδα μας. Του δίνουμε μεγάλη σημασία. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι στις τροπολογίες του κ. Ρούμπικ βλέπω δύο πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα είναι τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, πρέπει να το στηρίξουμε. Και κάτι που θα σας αρέσει, Πρόεδρε, γιατί εδώ και χρόνια εσείς αγωνίζεστε για ένα νέρασμο για ασκούμενους. Εδώ λοιπόν προτείνεται ένα έρασμος για νέους επιχειρηματίες. Οπότε μπορεί κάλλιστα να συμπεριληφθεί και αυτή η πτυχή στη γνωμοδότηση. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις του κύριου Ρούμπικ. Ευχαριστούμε κύριε Ντεπρέλη, ο πρόεδρος άλλος που θέλει το λόγο. Εγώ πρέπει να πω ότι φυσικά και χαίρομαι πάρα πολύ που απευθύνεται στους νέους επιχειρηματίες το Εράσμους. Το πιλωτικό πρόγραμμα, μάλλον μεταξύ των πολιτικών προγραμμάτων που κρίναμε σήμερα το πρωί, ένα από αυτά έχει να κάνει με το Makers. Είναι μια εμπειρία που έχουμε από τις ΗΠΑ, ε, δοκιμάστηκε στο MIT. Πρόκειται για νέους φοιτητές, μηχανικούς, οι οποίοι έχουν ένα σχέδιο στο μυαλό τους και θέλουν να το υλοποιήσουν. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζονται πολύ ειδικό εξοπλισμό για τρισδιάστατε, αντίγραφα κλπ. Άρα θέλουμε ε, με τις υποτροφίες αυτές του Εράσμους να τους επιτρέψουμε τρεις ή και έξι μήνες να μετακινηθούν για να υλοποιήσουν, να κάνουν συγκεκριμένο το σχέδιό τους. Αυτή είναι λοιπόν η ιδέα του makers, αυτών που κάνουν, που πράττουν. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την Επιτροπή Προπολισμών που σήμερα το πρωί ανέκρινε τα πιλωτικά αυτά προγράμματα. Μεταξύ άλλων και αυτό που όντως εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κύριε Ρούμπικ για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Καταρχά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη και σε ό,τι αφορά ε, την εγγραφή των ποσών ε, συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω το Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να συνδιαμορφώνει ενεργά το πρόγραμμα και να είναι όσο γίνεται λιγότερες οι δαπάνες που δεν έχουν ε, συγκεκριμένη αναφορά. Ε, ποιο χρονοδιάγραμμα έχει στο μυαλό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό τον καιρό, θα μπορούσε να μας πει. Alors, Monsieur ε, βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ρέλ. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, κύριε Ρουμπίκ, αλλά ευχαρίστως να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψε κολουφερών μεταξύ σας και θα μεταφέρω τις ερωτήσεις σας. Πρόεδρος. Ωραία, το αφήνουμε εδώ λοιπόν το θέμα και διευκρινίζουμε ότι οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 6 το απόγευμα στις 10 Οκτωβρίου και ότι η Επιτροπή Προπολογισμών στις ε, 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσει. Τώρα, κυρία Γκαρτζιά Θαμπάλ, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Θάλασσας και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τηλεγραφικά. Έχουμε τρεις ε, γραμμές εδώ στη γνωμοδότηση. Το ένα είναι να ε, τονίσουμε εκ νέου τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι ε, πολύ κοντά σε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα Δεύτερον, να σεβαστούμε τα νούμερα του σημερινού δημοσιονομικού πλαισίου και σεβόμενοι αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, συνομιλώντας με τους αρμόδιους της Επιτροπής Αλίας, θεωρήσαμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει λίγο πιο πέρα από τους στόχους που είχαμε μέχρι τώρα στο Ταμείο Θάλασσας και Ελίας. Επομένως, ε, για να ε, μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους νέους ε, στόχους και να οδεύσουμε προς την γαλάζια οικονομία, είπαμε ότι θέλουμε μία αύξηση 10%. Και η τρίτη πρόταση είναι ότι καθώς ε, ως κοινοβούλιο αυξάνουμε τις δαπάνες για την κλιματική αλλαγή στο 30% σε αυτό το τομείο, το οποίο συνδέεται ιδιαίτερα με το θέμα, περνάμε το 30% στο 35% για να αντισταθμίσουμε άλλα ταμεία που δεν θα φτάσουν στο ποσό αυτό και να μπορέσουμε να έχουμε επομένως 30% συνολικά. Έτσι λοιπόν, στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, ε, συν 10% κονδύλια για τη υλοποίηση των στόχων και 35% για το κλίμα. Ευχαριστώ. Έιντερ. Σκιώδης, ε, σκιώδης εισηγήτης. Μέσω του κύριου Βερδάντης, ο κ. Γκοτσάλες ε, Πόνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω πορτογαλικά. Όχι, ισπανικά. Αλλά θα προσπαθήσω στα πορτογαλικά να αντικαταστήσω τον Ισπανό συνάδελφο. Ο συνόδελφος και ο δισηγητής του ΕΛΚ δεν μπορεί να είναι παρόν. Ζητώ συγγνώμη εξ ονοματός του. Ευχαριστεί την ε, εισηγήτρια για το έργο της και για την έκθεση. Συμφωνεί με τις ανησυχίες της και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την περικοπή που προτείνεται για μία από τις λίγες πολιτικές που, όπου έχει αποκλειστεί και αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα είναι ζωτικό θέμα επίσης και η σύνδεση με τη γαλάζια οικονομία. Και σύμφωνα με το στόχο που έχουμε να προωθούμε τις ε, βασικές πολιτικές. Ο εισηγητής συμφωνεί ότι αυτό είναι ένα ταμείο όπου οι περικοπές που προτείνει από την Κομισιόν είναι απαράδεκτες. Και είναι βέβαιος ότι η καλή συνεργασία με την εισηγήτρια θα οδηγήσει σε, μια καρποφόρο, σε ένα καρποφόρο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν την άποψη του κυρίου Γκονσάλε Πόνς μέσω του κυρίου Φερνάντε. Ο κύριο Τόρβαλτ έχει εξουσιοδοτήσει τον κύριο Ντεπρέ. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, αναλαμβάνω. Ευχαριστώ τη συνάδελφο. Βλέποντας τις τροπολογίες, αν μιλάμε για την αλία. γιατί σχεδόν το σύνολο των τροπολογιών μιλούν για στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια μιλάμε για την ισότητα των δύο φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της Ένωσης. Μετά μιλάμε για την αναγκαιότητα να πετύχουμε τους στόχους της COP21. Τους ε, συνεπογράφω, συμφωνώ με αυτούς τους γενικούς στόχους ε, όμως για την τελευταία πρόταση, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά, θα συζητήσω με τους συναδέλφους να δω ποια θα είναι η δική μας στάση και ίσως καταθέσουμε και τροπολογία. κύριος Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ ε, την εισηγήτρια θερμότατα. Ίντερ, είναι πολύ καλή η εκθεσευτή. Γιατί ακριβώ η γαλάζια οικονομία στο μέλλον θα παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Τα δύο τρίτα τη γης καλύπτεται από νερό. Ε, ε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ε, θέλουμε με τους στόχους αυτούς να έχουμε καθαρές θάλασσες και καλό περιβάλλον για τη διαβίωση και των ανθρώπων. Θα πρέπει οι ωκεανοί μας λοιπόν να απελευθερωθούν και να καθαρίσουν. Ερωτώ, σε αυτό το πρόγραμμα προβλέπετε και τίποτα για ε, τα πλαστικά απόβλητα στη θάλασσα ή διάφορα δίχτυα αλλιευτικά που ε, έχουν παρασυρθεί από τα νερά. Γιατί ξέρουμε που είναι η μεγαλύτερη ρήπανση των ωκεανών. Μπορούμε να το δούμε και με το Γαλιλαίο, με τα δορυφανικά προγράμματα, ε, ακριβώς να ε, εντοπίσουμε τα μέρη εκείνα στους ωκεανούς που έχουν μεγαλύτερη ρήπανση και στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας να βγάλουμε αυτό το πλαστικό, να το επεξεργαστούμε, να το ανακυκλώσουμε και ε, αφού μιλάμε και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είναι και προτεραιότητα, θα πρέπει οπωσδήποτε στο πρόγραμμα του το δω να ασχοληθούμε και με τους ωκεανούς που θα πρέπει να είναι και για τα ψάρια, όχι για τα πλαστικά. Ευχαριστούμε κύριε Ρούμπιχ. Κυρία Γκαρδία Σεμπάλ, με συγχωρείτε κυρία Τομά. Ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να συγχαρώ την συγκεντρία. Να προσθέσω κάτι. Το αίτημα του 10% το επενούμε και ανταποκρίνεται σε αυτές τις αρμοδιότητες, σε αυτούς τους νέους στόχους που έχουν να κάνουν με την καλαζή οικονομία. Όμως το 10% για την καλαζή οικονομία στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγο. Κυρίως ε, όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα που ξέρουμε ούτω ή άλλω ότι είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα διαφορετικά τομεία. Δηλαδή αυτό το 10% τα κονδύλια αυτά απλώς ε, θα χρησιμεύσουν για μελέτες. Γιατί βάσει και όσων υπόθηκαν προηγουμένως, το πρόβλημα των ωκεανών είναι ότι έχουμε ανεπαρκή δεδομένα για να αναπτύξουμε τη γαλάζια οικονομία είτε για να διασφαλίσουμε μία ε, ανάπτυξή της ε, ικανή, αλλά να προσθέσω και κάτι ακόμη για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη όχι μόνο η Αλία είναι μία από τις ε, πιο ολοκληρωμένες πολιτικές της Ένωσης, αλλά είναι αυτή που σχετίζεται περισσότερο με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή, κάθε κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την οικονομική ανάπτυξη, ακριβώς λαμβάνει υπόψη το σεβασμό των πόρων και των ωκεανών. Πρόκειται λοιπόν μια παραδειγματική πολιτική που θα άξιζε περισσότερα από δημοσιονομική σκοπιάς επίσης να πω ότι για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι έχουμε νέες αρμιδιότητες και νέους στόχους, μειώνοντας ταυτόχρονα τον προϋπολογισμό. Και ε, ακριβώς την κατηγορήσει αυτό πολύ καλά αυτή η έκθεση. Μάλιστα, κοιτάξτε τώρα η Σοφία είναι να ξέρει κανείς να μειώνει τον προϋπολογισμό. Ε, αυτό είπατε. Και εγώ το προσπεγράφω. Γιατί συλλογικά έχουμε το καθήκον ε, να ελέγχουμε τις δημοσίες δαπάνες. Και ελεγχθέν αυτών η συγγήτρια για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν, σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Να δώσω κάποιες απαντήσεις ε, στις αμφιβολίες του κ. Ντεπρέ ή στην έκπληξή του που μίλησα τόσο για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, για τις γυναίκες και για τους κλιματικούς στόχους στην εκθεσία αυτή. Ο τομέας της αλίας πιθανότατα είναι ένα από τους κλάδους όπου έχουμε μεγαλύτερη ανισότητα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά. Γι' αυτό ήθελα να το τονίσω σε αυτή τη γνωμοδότηση, σε ό,τι αφορά το κλίμα. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν θα έχουμε το 20% των δαπανών για το κλίμα, 5% και κατόπιν θα έχουμε μία συγκεκριμένη πρόταση και πρότειναν το 30%. Εμείς ως κοινοβουλίου ζητήσαμε το 30%, ανέβηκα στο 35% στην ειδική συμμετοχή αυτού του Ταμείου. Απλώς σε αυτό συνίσταται, αλλά αν έχετε άλλες προτάσεις ευχαρίστως να τις μελετήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Υπό τη μορφή τροπολογιών που πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα τις εξετάσει και θα τις ψηφίσει. Τώρα θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο Βόλκεν για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ναι, ευχαριστώ πολύ αξιότιμε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και πλέον και μπορούν εθελοντικά να υπηρετούν και να προσφέρουν οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασίζεται και στηρίζεται σε αυτή την ε, ε, επιτυχία του και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλε 100.000 νέου σε έξι διαφορετικού τομεί πολιτική να δραστηριοποιηθούν. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα. Στη γνωμοδότησή μου τονίζω και αλλάζω κυρίω τρία πράγματα. Πρώτον, και εγώ έχω δώσει τα ποσά σε σταθερέ τιμέ και όχι τρέχουσε, ε, όχι, δηλαδή constant και current prices. Ε, επίσης, ε, προτείνω το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συμμετέχει στην άρση των διακρίσεων και να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης του για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και υποστηρίζω ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων στην επιλογή των συμμετεχόντων εκεί εθελοντών και ένα τρίτο που έχω συμφωνήσει και, και ευθυγραμμίσει στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη θέλεις θέλησα να προσαρμόσω τους στόχους μας αυτά. Ελπίζω να μην ξανασυζητηθεί εδώ το θέμα του redeployment, όπως την περασμένη εβδομάδα ή την προπερασμένη στο Στρασβούργο. Καταφέραμε με κόπο μέχρι το 2021 να βρούμε χρήματα. Μην μας πάρουν τους πόρους τώρα από εκεί και τους ε, αφιερώσουν κάπου αλλού. και ελπίζω για τη νέα περίοδο 21 με 27 να ε, έχουμε ένα νέο πρόγραμμα χωρίς περιορισμούς και στενούς κορσέδες. Και τώρα με χαρά περιμένω την ανταλλαγή απόψεων ε, ε, του πλήθους των σχεδόν εισηγητών που παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Σχόλια από τον κύριο Νόβακοφ, μέσω του κύριου Φερνάντε όμω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Νόβακοφ είναι σε άλλη συνεδρίαση και δεν μπορεί να βγει στη Ρέγγι. Και ευχαριστεί για την έκθεση, ευχαριστεί τον εισηγητή κυρίω και λέει ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική για να προωθήσουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης και για την ε, μαθητεία, για την πολυπολιτισμική διάσταση. Είναι επίσης ένα πρόγραμμα μέσω το οποίο μπορούμε να προωθήσουμε τη γενοδορία και την αλληλεγγύη. Είναι πάντα στην ίδια γραμμή, όπως και το πρόγραμμα Erasmus ΣΥΝ. Πώς θα γνωρίσουμε τον άλλον. Πώς θα γνωρίσουμε τον κόσμο του. Μπορεί να αποτελεί στόχο για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Έτσι ώστε ο καθένας μας και οι δύο νέοι να νιώθουν πραγματικά Ευρωπαίοι με κοινέ αρχές στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πνεύματος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ μιλάτε υπέρ των νέων ώστε να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. κύριε, κυρία σίγουρα ζήτησε από τον κύριο Ντεπρέ να μιλήσει εκ μέρου τη. Σωστά τα λέτε, Πρόεδρε. Πρώτον, συμφωνώ απόλυτα με τους προσανατολισμούς που μας παρουσίασε ο κύριος Φερνάντες και φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούν Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα με τις τροπολογίες του εισηγητή, τον οποίο και ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία, άλλος κανείς. Έχει να προσθέσει τίποτα έτσι, ποιητικό άλλο. Κύριε Σίτα, νομίζω ότι ενθουσιάσατε την Επιτροπή Προπολογισμών. Α, ο κύριος Σόβαλτό όμως έχει το λόγο. Πολύ μου αρέσει πώς λέτε το όνομά μου, πώς το προφέρετε. Πρόεδρε, μια που έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να πω κάτι πολιτικό όσον αφορά τα προγράμματα αθελοντισμού και τα συναφή. Πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία. Πιστεύω ότι προσφέρουν στους νέους μια εμπειρία που δύσκολα θα την πάρουν αλλιώς. Αυτό όμως που με απασχολεί είναι ότι τα προγράμματα αυτά τελικά δεν αποδεικνύονται να είναι όπως ακριβώς θα θέλαμε. Ε, Κάποιο από το δικό μου το υπόβαθρο δεν θα έχει την ευκαιρία ποτέ να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα σαν κι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τα προγράμματα αυτά να μην είναι, οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην περιορίζεται μόνο στην μεσαία ευρωπαϊκή τάξη. Γιατί δεν είναι εκεί που υπάρχει το πρόβλημα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Έπειτα είναι χάσιμο χρόνου και χρήματος. Αυτά τα προγράμματα ελπίζω ότι όντως θα είναι επιτυχή, αλλά και να υπάρξει κοινωνικό μείγμα, να φροντίσουμε γι' αυτό. Να φροντίσουμε δηλαδή να γίνει σωστή δουλειά, ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα. Δηλαδή σε αυτά τα προγράμματα να αντικατοπτρίζεται η σύνθεση της ευρωπαϊκής κοινωνίας και κοινωνικά όσον αφορά τις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε κύριε Χάουαρτ. Ωραία. Για να ολοκληρώσει ο κύριος Βόλκερ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα όσα είπε μόλις ο πρόλαλής σας. Επιστεύω πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό πραγματικά καλύπτει όλο το φάσμα των νέων στην Ευρώπη και μπορεί να το κάνει. Ε, είναι πάρα πολύ ανοιχτό, αφορά περιόδους άσκησης, μαθητείας σε διάφορους τομείς, ε, εθελοντική προσφορά. Είναι πάρα πολύ τομείς, πραγματικά. Και έτσι πιστεύω και εγώ ότι το πρόγραμμα αυτό είναι το κατεξοχήν πρόγραμμα που δημιουργεί ε, αυτό, φτάνει σε αυτό το στόχο που έχει, δηλαδή να ε, φτάνει σε ευρεία στρώματα, ευρεία στρώματα της κοινωνίας. Ε, χαίρομαι που έχετε θετική εικόνα για το πρόγραμμα και γνωμοδοτείτε θετικά. Ευχαριστώ. Σίγουρα ε, συμφωνούν όλοι. Εάν υπάρχουν τροπολογίες, παρακαλώ να κατατεθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Εμείς θα ψηφίσουμε εδώ στις 5 Νοεμβρίου. Και τελειώνει εδώ αυτή η ωραία συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν έχετε τίποτα στα διάφορα να θέσετε. Όχι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, 8 και 9 Οκτωβρίου θα συνεδριάσουμε στις Βρυξέλλες, θυμίζω. 22 Οκτωβρίου θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών στο Στρασβούργο, όπως και στις 25 Οκτωβρίου και άλλη κοινή συνεδρίαση Badge Econ στο Στρασβούργο. Φτάνουμε λοιπόν στο πέρας ε, αυτής της εβδομάδας που είναι η πιο επίφοβη για την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών, γιατί εξετάζουμε όλες τις τροπολογίες του προϋπολογισμού για να αποκρισταλώσουμε το σχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Φέτος επιβαρύνθηκε αυτή η δοκιμασία από το γεγονός ότι έπρεπε να αποφανθούμε και για σχέδια γνωμοδότησης, για προγράμματα του πολιτούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. 27 παρακαλώ προγράμματα εξετάσαμε αυτό το τριήμερο. Εκτός από την κλασική δημοσιονομική διαδικασία. Μπορεί να μην το πήρατε είδηση, αλλά όλοι οι συνεργάτες μας και οι υπάλληλοι ε, μια τεράστια πίεση, αλλά έκαναν και καταπληκτική δουλειά. Και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους εκ βάθους καρδίας για τον επαγγελματισμό τους και την απόλυτη αφοσίωσή τους, την ευφία, την ενέργειά τους και την μόνιμη αισιοδοξία τους, όπως και εμείς πιστεύουν και εκείνοι στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ και τους πολιτικούς συμβούλους και υπαλλήλου των διαφόρων πολιτικών ομάδων, όπως και όλους εσάς συναδέλφοι, Ιδιαίτερα τους, τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Αυτά. Λήξη συνεδρίασης. Ε, καλό υπόλοιπο εβδομάδας και καλό Σαββατοκύριακο.